Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μα. Έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Προτείνονται οι εξή αλλαγέ στο σχέδιο ημερήσια διάταξη. Αναβάλλεται το σημείο 12. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται το σχέδιο ε, ημερήσια διάταξης με αυτή την τροποποίηση. Η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά από το ίντερνετ και ότι οι χρόνοι που προβλέπονται για κάποιο θέμα είναι απλώς ενδεικτικοί και μπορεί να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Το σημείο 3. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Να σας ενημερώσω ότι οι συντονιστές στη συνεδρίασή τους της 20 Νοεμβρίου αποφάσισαν τα εξή. Πρώτον, να καλέσουν την Επιτροπή να παρουσιάσει την ανακοίνωσή της για τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις μας πριν από το τέλος της θητείας. Δεύτερον, να στείλουμε μία απάντηση στην Ένωση Πρώην Μελών για το πρόγραμμα συντάξεων των μελών και μια απάντηση στην επιστολή για το αίτημα άρσης ασυλίας ενός μέλους. Επίσης αποφάσισαν για τη διαδικασία του, του, της πρότασης ψηφίσματος για το UPCA. Αποφάσισαν ότι οι γνωμοδοτήσεις για μια συνολική ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και την ρομποτική ε, για την Ήτρε και η γνωμοδότηση για την τροποδότηση του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την ε, ΑΦΧΟ θα αποσταλούν μέσω επιστολής. Αποφάσισαν να υπάρξει μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 10 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Να ορίσουν τον κύριο Χρυσόγωνο ως εισηγητή για την αίτηση άρσης ασυλίας ε, του Ζώμα Ιλουπέν και μέσω σωρατής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε στις 27 Νοεμβρίου οι συντονιστές αποφάσισαν επίσης να ορίσουν τον κύριο Χρυσόγονο ως εισηγητή για την άρση ασυλίας της κυρίας Ντομινίκ Μπίλντα. Τώρα, στη σημερινή μας συνεδρίαση οι συντονιστές αποφάσισαν να ορίσουν την κυρία Μπερζό η συγκίτρια γνωμοδότησης για το σχέδιο συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ του Eurojust και της Γεωργίας. Επίσης, ορίστησαν μόνιμοι εισηγητές για την νομική βάση, ο κύριος Λιποετών, για την επικουρικότητα, ο κύριος Τζαμπάσκι για επίμαχα θέματα, η κυρία Φεράρα, για την επιτροπολογία, ο κύριος Καβαντά, και για την κωδικοποίηση και τις αναδιατυπώσεις, ο εισηγητής θα είναι ο κύριος Χρυσόγονος. Επίσης. Ετήματα άρσης ασυλίας. Κοινή αντιμετώπιση για τους κυρίους Φουντούλη, Συναδεινό και Επιτίδιο. Θα τον αναλάβει ο κύριος Τζαμπάσκη. Και στην περίπτωση του κυρίου Ντόρμαν θα είναι η συγκήτρια η κυρία Ρέγναρ. για την περτέρω πρόοδο όσον αφορά το θέμα κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο αποφασίσαμε να στείλουμε ένα γράμμα στην Επιτροπή Προέδρων Επιτροπών και τέλος οι συντονιστές συμφώνησαν να αποσταλεί επιστολή στον πρόεδρο της ΑΦΚΟ όπου διαμαρτυρόμεθα για τη διαδικασία για τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια των ε, ευρωεκλογών. Αυτές ήσαν οι ανακοινώσεις. Τέσσερα. Επικορικότητα. Δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε περνάμε στο 5. Εξέταση του σχέδιου εκθέσεως για τη δράση της Ένωσης μετά την ε, ένταξή της στην ε, πράξη της Γενέβης ε, της Συμφωνίας της Λισαβόνας για ονομασίες προέλευσης και βιογραφικές ενδείξεις. Και να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Γοζιέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπογραμμίζω ότι η πρόταση κειμένου αυτή υπάρχουν δύο μέρε. Υπάρχει μία σύμφωνη γνώμη σε μία απόφαση του Συμβουλίου για να ενταχθούμε στην πράξη της Γενέβης και μια πρόταση κανονισμού που έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε ως Κοινοβούλιο. Υπογραμμίζω ότι το κείμενο που έχουμε ενώπιόν μας μου δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ θετική η επιτυχία αυτή της Ένωσης, ούτω ώστε να προστατεύουμε τις γεωγραφικές μας ενδείξεις. Η διπλωματική συνδιάσκεψη του 2015 που κατέληξε στην έγκριση της πράξης Γενέβης και που επιτρέπει στην Ένωση να συμμετέχει στη διευθέτηση της Λισαβόνας είναι καλή είδηση για τους Ευρωπαίους παραγωγούς που μέσω αυτής της συμφωνίας θα ωφεληθούν στα πλαίσια των διεθνών συναλλαγών η ιδιαιτερότητα των προϊόντων τους θα προστατεύεται και έχουμε μια μακρά παράδοση προστασίας τοπικών προϊόντων. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που όντως ε, θα λάμψουμε στο διεθνές εμπόριο χάρη σε αυτή τη συμφωνία. Ωστόσο, η αρχή αυτή, ε, η πρόταση αυτή μου δημιουργεί διάφορες ανησυχίες. Πρώτα απ' όλα ο κατάλογος των γεωγραφικών ενδείξεων που θα γνωστοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την ένταξη σε αυτή την πράξη της Ένωσης. Η Επιτροπή στην πρότασή της. λαμβάνει το δικαίωμα, σφετερίζεται το δικαίωμα να ορίσει ε, ποιες είναι οι γεωγραφικές ενδείξεις που θα πρέπει να προστατεύονται. Δεν είναι αυτή η σωστή λύση. Πρέπει να επιστρέψουμε στους παραγωγούς επιτόπου. Αυτοί γνωρίζουν την πραγματικότητα της ε, δράσης τους, της παραγωγής τους, των αγορών τους, ε, τον, ε, ε, εκεί που διαθέτουν τα προϊόντα τους. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί να υποβάλουν τα αιτήματα για αναγνώριση γεωγραφικών ενδείξεων. Και τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να έχουν το ρόλο τους. Γιατί τα κράτη-μέλη εποπτεύουν και ε, δημιουργούν τους οργανισμούς διαχείρισης που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση ακριβώς των γεωγραφικών ενδείξεων. Όπως θα δείτε λοιπόν, τροποποίησα προς αυτή την κατεύθυνση το κείμενο ούτω ώστε να μπορέσουν να παρέμβουν όντω οι παραγωγοί και όλοι όσοι παρεμβαίνουν επί τόπου. Και εκεί που έχω τα περισσότερα προβλήματα και εκεί που είμαι ιδιαίτερα απογοητευμένοι είναι ότι η πρόταση αυτή δεν συνοδεύεται από ένα μηχανισμό προστασία των υγραφικών ενδείξεων για τα μη γεωργικά προϊόντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ξέρουμε πολύ καλά, εμεί εδώ ιδιαίτερα ω Επιτροπή, ότι υπάρχει αναγκαιότητα για κάτι τέτοιο να το θέσω στο πλαίσιο. Η συμφωνία τη Γενέβη επιτρέπει να προστατεύουμε και οι γεωγραφικέ ενδείξει για μη γεωργικά προϊόντα. Αυτό μα προσφέρεται μέσω αυτή τη πράξη. Αλλά επειδή η Ένωση σήμερα εξακολουθεί να μην έχει νομοθεσία για τα θέματα προστασία μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων, μα προτείνει η Επιτροπή ένα κείμενο που δεν μα επιτρέπει να υπάρξει διεθνή αναγνώριση για αυτά τα προϊόντα. Και αυτό είναι απόλυτα παράδεκτο, κατά τη γνώμη μου. Το 2013 για να επενθυμίσω στη συζήτηση που κάναμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια μελέτη πολύ πλήρη που κατέληξε ότι υπάρχει αναγκαιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ωφεληθεί μέσω νομοθεσίας για τις μη, γεωργικ... μη γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις. Το 2016 εγώ ήμουν εισηγήτρια μιας έκθεσης που ε, εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2016 συγκεκριμένα με πολύ ευρία πλειοψηφία από την Επιτροπή μας και από την ε, Ολομέλεια όπου καλούσα να ε, δοθεί συνέχεια σε αυτά που είχαμε ήδη αποφασίσει αλλά έκτοτε δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει αντίθεση αρχής, δεν ξέρω τι είναι, αδράνεια. Τίποτα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν προστατεύονται οι μη γεωργικές, γεωγραφικές ενδείξεις. Ε, κάτι όμως που, για το οποίο καλούν ε, τα κράτη-μέλη, η τοπική αυτοδιοίκηση, όλα τα επιμελητήρια, το κοινοβούλιο, επαγγελματικέ ενώσεις, τα πάντα. Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Η πράξη αυτή ε, λοιπόν θα έχει πολύ αρνητικέ επιπτώσεις. Γιατί μία αρμοδιότητα που έχουμε και είναι αναγκαίο να την μεταφέρουμε βεβαίω. Γιατί εμείς έχουμε την ε, αρμοδιότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, για την προστασία των γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων, αλλά επειδή έχει υπάρξει ανα, αδράνεια από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να, ε, να κινητοποιήσουν, να ενεργοποιήσουν καλύτερα αυτήν την ε, προστασία των μη γεωργικών ε, γεωγραφικών ενδείξεων. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει καμία πλέον δυνατότητα να προστατεύσει αυτές τις γεωγραφικές ενδείξεις. Άρα θα υπάρξει στην ουσία πισωγύρισμα αυτή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα αρνητική και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο εάν ταχαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα οριζόντιο κείμενο για να προστατεύσει και τι μη γεωγραφικέ ενδείξει για να ενταχθούμε πλήρω στην πράξη τη Γενέβη. και οι τροπολογίε που υπέβαλα αυτό προσπαθούν ούτω ώστε στο τέλο να υπάρξει ευρωπαϊκή προστασία για τι μη γεωργικές ενδείξει. Θα ζητήσουμε λοιπόν εγγυήσει από την Κομισιόν δεν μπορεί να περάσει αυτή η πράξη χωρί να λάβει σαφή θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επέκταση και στι μη ε, γεωργικέ ενδείξει. Και είναι προπόθεση αυτό για να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μα για να ενταχθεί η Ένωση στη πράξη τη Γενέβη. Αδειμονώ λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με του συναδέλφου και ελπίζω να υπάρξει η ίδια δυναμική και η ίδια ομοφωνία που υπήρξε και το 2016 για τις γεωργικές ενδείξεις για να προστατεύσουμε επιτέλους πλήρω το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Τεχνογνωσία. Ευχαριστώ κύριο Καβαντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ πλήρω με την πρόταση της κυρίας Γοζιέ και είναι ανησυχητικό το ότι η Κομισιόν δεν εγγυάται οριζόντια προστασία. Πρέπει να ολοκληρώσει την εργασία της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρέπει λοιπόν να διορθώσει την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απευθύνω έκκληση προς αυτήν ταχαίω. Ταχύτατα. Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πει τίποτα. Σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε Είμαι ο Κλάου Μπλάνκ από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Για 20 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί επιτυχή πολιτική προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και στη διεθνή αγορά και σε τρίτες χώρες. Η πολιτική αυτή ωφελεί σαφώς ε, τους παραγωγούς και δημιουργεί απασχόληση και ανάπτυξη. Έχουμε κάνει πολλέ προσπάθειες και πολιτικό κεφάλαιο για να θεωρηθεί η Συμφωνία τη Λισαβόνα. Η Ένωση τώρα πρέπει να εφαρμόσει την ισχύουσα πολιτική της και να ε, ενταχθεί στην πράξη της Γενέβης είναι σημαντικό να υπάρξει ταχεία πρόοδος για να λειτουργήσει σωστά η ενιαία αγορά και για το Διεθνές Θεματολόγιο για την προστασία των ενδείξεων ε, που έχει η Ένωση. Αυτή είναι η καλύτερη και η μόνη νομικά βάσιμη προσέγγιση. Δεν θα πρέπει να δημιουργεί αμφιβολίες ε, στους παραγωγούς που θα ωφελούνται στην ε, εξαγωγή των προϊόντων τους σε τρίτες χώρες και δεν θα έχουν μειονεκτήματα. Και βεβαίω είναι αποκλειστική αρμοδιότητα, η, η Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά. Χωρί να προκαταλαμβάνω την επίσημη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια τη κανονική ε, νομοθετική διαδικασία, να κάνω κάποια σχόλια για τι ε, προταθήσει τροπολογίε. Πρώτον, σημειώνω ότι υπάρχει από ό,τι φαίνεται ομοφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή, για το στόχο τη επιτυχού και ταχεία ένταξης της Ένωση στην πράξη της Γενέβης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί η ταχεία ένταξη θα είναι κρίσιμη για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος Λισαβόνα λόγω της απόλυτη εχθρότητα προς το σύστημα αυτό που επιδεικνύουν σημαντικά μέλη του ΠΟΕ και ιδιαίτερα οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά για να υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί εγκαίρω αυτό ο στόχο δηλαδή μέσα στον επόμενο χρόνο και ελπίζουμε με πριν από την, ε, προηγούμενη, την επόμενη Γενική Συνέλευση του ΠΟΕ δεν πρέπει να ε, ξεχνάμε το γενικότερο νομικό και πολιτικό πλαίσιο. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες λοιπόν, γιατί κάποιες από τις τροπολογίες που προτείνονται στο κείμενο της εισηγήτριας δεν βελτιώνουν τον κανονισμό. Αλλά επιπλέον μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην ε, έγκρισή της. Ιδιαίτερα η τροπολογία 2, αιτιολογική σκέψη 4. Όπως λέει η τροπολογία 3 λοιπόν αναφέρει, ο ε, μεμονωμένος παραγωγός θα πρέπει να έχει λόγο μόνο σε ε, εξαιρετικές περιπτώσεις. Τροπολογία 6 για ένα, μια νέα αιτιολογική σκέψη 8α. Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει τέτοια δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να ενταχθούν στην πράξη της Γενέβης για να προστατεύσουν τις γεωγραφικές ενδείξεις που δεν έχουν οριζόντια προστασία σε ενωσιακό επίπεδο. Αυτό είναι το πιο προβληματικό θέμα από τις προτινόμενες τροπολογίες. Και η τροπολογία 9. Νέα αιτιολογική σκέψη 11b. Ναι μεν. Διαβεβαιώνω την Επιτροπή σας ότι έχουμε κάθε κατανόηση για τα αίτια υποβολής αυτής της τροπολογίας ε, θα ήθελα να σας πω ότι δεν νομίζω ότι είναι ε, το σωστό σημείο για να παρατηρήσει αυτό το θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν θέλουμε να επιτύχει αυτή η ένταξή μας στην πράξη της Γενέβης, η νομοθετική διαδικασία δεν θα πρέπει να περιπλακεί με το θέμα της νομοθεσίας για τις μη γεωργικές ενδείξεις. Είναι χωριστό θέμα. Η πρόταση της Επιτροπής έχει διατυπωθεί πολύ προσεκτικά για το θέμα αυτό δεν επηρεάζει ούτε προκαταλαμβάνει το θέμα ε, εάν και κατά πόσο θα πρέπει να εγκριθεί ενωσιακή νομοθεσία για μη γεωργικέ ενδείξει. και αυτό επειδή αναγνωρίζουμε την νομική και πολιτική πραγματικότητα. Αυτό είναι το πιο προβληματικό θέμα. Τονίζω, υπάρχει κίνδυνος να εκτροχιάσει τη διαδικασία ένταξη τη Ένωση. Τώρα τροπολογία 10, άρθρο 2.2. Έχω μια ερώτηση. Μήπως η συγκήτρια μπορεί να επιβεβαιώσει ότι είναι σορευτικές οι προϋποθέσεις. Δηλαδή όλες αυτές οι ενδείξεις που τώρα ωφελούνται από αυτή την προστασία και είναι στο Διεθνές Μητρό ε, τις έχουν εντάξει, δηλαδή τα κράτη-μέλη που είναι μέλη ήδη αυτή τη πράξη ε, τις έχουν εντάξει σε αυτό το διεθνέ μητρό. Τροπολογία 12. Για το άρθρο 2-3. Ε, με συγχωρείτε κύριε. Μπορείτε να τελειώνετε. Οπότε συνοψίζω, λέει ο πρόσωπο Κομισιόν. Ποιο είναι το πιο προβληματικό θέμα. Αυτή η εστίαση στι μη γεωργικέ ε, ενδείξει. Και ιδιαίτερα στην τροπολογία 18 που ε, εκφράζει ανησυχίε ε, συστημικού χαρακτήρα για το δικαίωμα πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ολοκληρώνω. Οι υπηρεσίε τη Κομισιόν είναι στη διάθεση του Κοινοβουλίου για υποφελή διάλογο και συνεργασία για τα θέματα αυτά με στόχο να διασφαλίσουμε την επιτυχή ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας και κατά συνέπεια να υπάρξει ταχεία ένταξη στο σύστημα της Λισαβόνας της Ένωσης ε, προς το συμφέρον των παραγωγών και άλλων εμπλεκομένων. Πολύ σύντομα. Θα αναφερθώ σε αυτό που είπε ο Μποσιέ, καθότι είμαι υπέρ του κοσμικού χαρακτήρα θα ήθελα πραγματικά να πω ότι πολλές φορές ε, εδώ ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέτα. Βεβαίως η πρόθεση της Επιτροπής είναι καλή, σε καμία όμως περίπτωση εδώ δεν υπάρχει αποτελεσματική δράση και οι αιτίε αυτού που προκάλεσε η δράση της δεν έχει καθόλου αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ. Στις 12 Δεκεμβρίου το μεσημέρι είναι η προθεσμή, την υποβολή α, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρο του 17 Δεκεμβρίου. Στις 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμή για την υποβολή τροπολογιών. Έχω ακόμα ένα σημείο, το σημείο 6, που είναι η ανταλλαγή απόψεων για το θέμα μιας ολοκληρωμένης ε, βιομηχανικής πολιτικής που αφορά την ε, τεχνητή νοημοθένη και την ρομποτική. Η κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, οι συντονιστές αποφάσισαν ότι η νομοδότησή μας για την έκθεση της Επιτροπής Ήτρε θα γίνει υπομορφή επιστολής. Εστάληχτε στο βράδυ αυτή η επιστολή αργά. Σε γενικές γραμμές υπενθυμίζουμε το ψήφισμα που υιοθετήθηκε με θέμα την ρομποτική καθώς και τα νομικά αποτελέσματα, τα νεοδουλικά αποτελέσματα του 2017 είναι αυτό το ψήφισμα. Λυπούμαστε πολύ γιατί καθυστέρησε η αντίδρασή μας. Βεβαίως και χρειάζεται μια συμμαχία από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα τεχνητής νοημοθύνης, να γίνει αξιολόγηση όσον αφορά τα προϊόντα που υπάρχουν, καθώς και όλο το δεοντολογικό κομμάτι αυτών των εφαρμογών. Βεβαίως και ο Αντιπρόεδρος θα υποβάλει ένα σχέδιο δράσης, ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής, ε, για την δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλή αργά παρά Περιμένουμε λοιπόν και θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων σε μία από τις πτυχές που είναι η τυποποίηση. Δεν την εξετάσαμε αρκετά, δεν την έχουμε καθόλου αν θέλετε, αναλύσει όσον αφορά τους ε, κανόνες και τα πρότυπα ISO. Προετοιμάζεται μια ολόκληρη σειρά προτύπων που θα αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προασπιστούμε εδώ τις αξίες μας αλλά και τις ε, δικές μας θέσεις σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, όσον αφορά το λεγόμενο fitness check, το θέμα της αντοχής της ε, η προσπάθεια αυτή θα πρέπει διαρκώς να ανανεώνεται. Όπως ξέρετε πρόκειται για μια τεχνολογία που εξελίσσεται με ταχύτητα τους ρυθμούς και είναι πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε πάντα ενημερωμένοι. Έχετε όλη την επιστολή αυτή, ελπίζω να την διαβάσετε, έχετε τη δυνατότητα να σχολιάσετε και να προσθέσετε, αλλά ο χρόνος είναι πολύ λίγος μέχρι αύριο το βράδυ. Πρόκειται για έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και φυσικά δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη όσον αφορά το αποτέλεσμα. Η Επιτροπή θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Βεβαίως και καλωσορίζουμε αυτήν την προσπάθειά σας. Θα υιοθετηθεί αύριο. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι των διοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών θα υπάρξει περαιτέρω διαβούλευση 18 Δεκεμβρίου. Thank ευχαριστώ. Νομίζω λοιπόν ότι ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Έχετε τόσο μεγάλους ε, καταλόγους πληροφορία. Μάλλον ο Άγιος Βασίλης μας τα άφησε γιατί έχουμε πολλά δώρα. Ο κύριος Άντερσον έχει ζητήσει το λόγο. Όχι. electronically? Everything. Everything? I mean, all the final votes. Yes. Okay, dear colleagues, are we prepared to vote? Είστε όλοι έτοιμοι, συνάδελφοι, για την ψηφοφορία. Έχετε τις κάρτες σας τη θέση τους όλοι. Okay, so we vote. Ξεκινάμε με την έκθεση Axel Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πρόκειται για το θέμα της βιωσιμότητας. Αρχή της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια κύριε Φως. Έκθεση Μπερζερό Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Αρχή της ψηφοφορίας Απορρίπτεται. Κυρία Μπερζερό, ξέρω ότι όταν απορρίπτεται μια έκθεση, μπορούμε να εξαλειφθεί το όνομα του εισηγητή. Εγώ ζητώ ακριβώς το αντίθετο. Θα ήθελα να υπογραμμιστεί το όνομά μου, να παραμείνει. Σας ευχαριστώ πολύ που την καταψηφίσατε. Θέλω να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου. Πρόεδρος. Περνάμε στο θέμα της ε, σύγκλησης, της διασυνοριακής, συγχωνεύσεις και διαιρέσεις. Περνάμε στην ε, 1. Α, συγγνώμη. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 252 υπέρ κατά. Μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. 2.46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 ονομαστική ψηφίζουμε και περνάμε στην συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6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 Περνάμε στην 13, συμβιβαστική 13, δεν υπάρχει 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 Έκανα λάθος. Η 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Ανα ελέγξουμε την 130. Η κυρία Ρέγνερ, ζητώ συγγνώμη πρόεδρε, νομίζω ότι ξεχάσαμε την Τροπολογία 496 της Πασκάλ Τυρό, του Πασκάλ Είναι ακριβώς πριν την ε, συμβιβαστική 13 και νομίζω την ξεχάσαμε. Πριν την 13 λέτε. 496 τροπολογία. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έκανα λάθος. Πρόκειται για το άρθρο 86. Παράγραφος 3. 4-9-6 είναι η τροπολογία υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Yes. And that's been adopted. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 629 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική Α, όχι. Έξι σαράντα εννέα υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την έξι εννέα. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην συμβιβαστική 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 44 α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάμε στην συμβιβαστική 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 49 υπέρ όχι 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 787 τροπολογία υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 787. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 61 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 ζητάτε ηλεκτρονικό έλεγχο 135 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 135 εγκρίνεται. ένα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η... Καταπίπτει η επόμενη. 136 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίνεται, θα έλεγα. Οίκον 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος του. Εγκρίνεται οι δύο. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 3 παρακαλώ. Εγκρίνεται η τρία, 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 4. Τα χέρια σας δεν είναι πολύ σαφή. Εγκρίνεται. 4, 140 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. 140 ελέγχουμε. Εγκρίνεται. Πέντε υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την πέντε. νομίζω εγκρίνεται 142 υπέρ κατά Να ξαναρχίσουμε. Θέλω να βλέπω τα χέρια σας. 142 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 144 καταπίπτει. 6 της οίκων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 147. Απορρίπτεται η 147. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά ελέγχουμε την 7 απορρίπτεται Τρία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την ε, τρία. Την τρία. Απορρίπτεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 153 και 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 154 και 5 υπέρ κατά να ελέγξουμε τις δύο προηγούμενες Ελέγχουμε την 153 και 152. Απορρίπτονται. 154 και 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 4 υπέρ. Να ελέγξουμε στην 4. Εγκρίνεται η τέσσερα. Πέντε, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την πέντε. 5. Απορρίπτεται. 155. 156 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται συμβιβαστική 62 εγκρίθηκε 162 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Απορρίπτεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 8. Εγκρίνεται, έκανα λάθος. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο για την 164. Ελέγχουμε. απορρίπτεται. Μια σειρά συμβαστικών ε, έχουν ε, εγκριθεί Περνάμε λοιπόν ε, στην ε, σκέψη 12α, τροπολογία 10, έμπλ, τροπολογία 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 12 έμπλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Αιτιολογική σκέψη 13-182 παρακαλώ. Ετυλογική σκέψη 16, 182, υπέρ. Ετυλογική σκέψη 16, 182, υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ετυλογική σκέψη 19α 16 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ. Δεν είμαι βεβαίως. Εγκρίθηκε. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 74. Στην εκλογική σκέψη 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 198. Προπολογία του κύριου Καρύμ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 77 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Οίκον 26 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 26 ήταν αυτή. 27 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 της υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 208 και 23 μαζί, 23 μαζί, υπέρ, κατά, άποχες, Εγκρίνεται. Η 209 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Παρακαλώ για τη 209. Απορρίπτεται. Η 210 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 90 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 91, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 92 υπέρ. Α, έχει εγκριθεί. Τροπολογία 216 στην ιδεολογική σκέψη 41 υπέρ. Κατά. Απόχες. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε για να είμαστε σίγουροι. Για τη 216 παρακαλώ ψηφίζουμε. Απορρίφθηκε. «25 της Επιτροπής Απασχόλησης. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 230. Ετυλογική σκέψη 48. 230. Υπέρ. Τι βρήκατε? Ετυλογική σκέψη 48, τροπολογία 230. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 231 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οίκον 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 107 για την αιτιολογική σκέψη 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 240 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 240. Απορρίπτεται. 241. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 242. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Απορρίφθηκε. 243 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 244 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικά τώρα την έκθεση του συνολό της παρακαλώ. Εγκρίθηκε. Και η απόφαση για έναξη των διαπραγματεύσεων. Μας λείπουν ακόμα τρία άτομα, τρεις ψήφοι. Και πέρασε τη ψηφοφορία τώρα. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Στην κυρία Ρέγνερ. Έχετε το λόγο, ναι. Εν συντομία, βλέπετε ότι υπάρχουν τόσε πολλέ συμβιβαστικέ προτάσει. Ήταν πραγματικά τεράστιο ο όγκο τη δουλειά. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ του κοιόδε συζητητέ, οι οποίοι μερών ε, δούλεψαν και ευχαριστούμε και το προσωπικό μας. Και αυτό αποτελεί και ένα σημάδι, μια ένταξη προς το Συμβούλιο. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε και αποτελεσματικά και γρήγορα και είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσει. Thank ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα έχουμε την έκθεση του κυρίου Ντιτιέ. για τις αντιπροσωπευτικές δράσεις. Ναι. Uh, Και να ξεκινήσουμε με τη συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Μετά έχουμε μια προφορική τροπολογία. Ως προσθήκη. Υπέρ. εξ ονόματο των Σοσιαλδημοκρατών. Σηκωθείτε παρακαλώ στην συνάδελφοι. Δεν συμφωνούμε με την προφορική τροπολογία. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρο. Άρα δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε, δεν είναι παραδεκτή. Και περνάμε στη συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική τρία Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Uh, uh, ναι, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Είχαμε ένα αίτημα της Γκουε για ονομαστική κλίση για όλες τις συμβιβαστικέ. Εξακολουθεί να ισχύει το αίτημά σας αυτό. Βεβαίω. Σας ζητώ συγγνώμη. Και άρα ξεκινάμε εξ αρχής πάλι. Συμβαστική 1. Ψηφίζουμε. Εγκρίθηκε με σαφή διαφορά. Συμβαστική 2. Ψηφίζουμε. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 3. Ψηφίζουμε. Εγκρίθηκε. Ήμκο 25. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. Ήμπκο 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ίδια μου φαίνεται η πλειοψηφία, αλλά θα λέξουμε παρακαλώ. Όχι. Αυτή εδώ εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 4 ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 5 τώρα. Ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε. Η 32 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 7. Ψηφίζουμε. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 479. «479, παρακαλώ υπέρ». «Κατά». «Έλεγχος». Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 7α, ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 8. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Ήμικο 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 454. Εγκρίθηκε. ΥΜΚΟ 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 456 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 457 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Απορρίπτεται. 458 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Σεμεβαστική 11. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 467. 467. υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 468. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 469. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 469. Απορρίπτεται. 470 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 471 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Συγγνώμη, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 488 ε, τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 41, ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε. 495 υπέρ. Κατά. Αποχές Έλεγχος παρακαλώ. Εγκρίθηκε. 497 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 536, τροπολογία 536. Στο παράδειγμα 1. 536, τροπολογία υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 67 και 538 από κοινού. Ψηφίζουμε. Περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 539 και ΙΜΚΟ 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ για την Ήμκο 64. Απορρίφθηκε. Η 541 και ΙΜΚΟ 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Γιατί είναι οριακό το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Μάλιστα. Απορρίπτεται. «542 και ΙΜΚΟ 68 υπέρ». Κατά. Η ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε αυτό το επιθυμείτε. Πέρας. «543 και ΙΜΚΟ 83 υπέρ» κατά αποχές νομίζω ότι η ίδια πλειοψηφία είναι αλλά αν θέλετε ελέγχουμε ελέγχουμε λοιπόν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Απορρίπτεται. Ήμκο 66. Υπέρ. Κατά. Την άλλη δεν καταλαβαίνω. Μάλιστα. Εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε. Λείπει μία ψήφος. Απορρίπτεται. 544 και ημικο 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 554 και 545. Υπέρ. Κατά απόχες απορρίπτεται 547 και 620 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 548 και ύμικο 71 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 549 και 71. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5.50 και ΙΜΚΟ 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Θέλετε να ελέγξουμε την 550 και την ΙΜΚΟ 72 ταυτόσιμες. Εγκρίθηκε. Συγγνώμη. Λάθος. 551 υπέρ. Κατά. Έλεγχο παρακαλώ. Μια ψήφος λείπει. Πέρασε. Εγκρίνεται. Πεντακόσια υπέρ. Συγγνώμη, ζητώ. 552 και ΙΜΚΟ 73 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Απορρίπτεται. 553 και 584 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 555 για την 25 υπέρ. Κατά. Απόχες. Έλεγχος. Αλλά έχουμε αυτές τις τρεις. 555, 556 και 75. Βλέπετε. Ισοψηφία και πάλι. Μάλιστα. Θέλετε να ψηφίσουμε και την επόμενη ηλεκτρονικά μήπως. Κατευθείαν. Α, την ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 557. Και οι υπόλοιπες. Απορρίπτεται. Λοιπόν, ηλεκτρονικά και για την 558 και ΙΜΚΟ 76. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 559 και 592 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Α, θέλετε έλεγχο. Καλός ηλεκτρονικός έλεγχος. Απορρίπτονται. 561 ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται.

Απορρίπτεται. 5.65. Απορρίπτεται. 604. Απορρίπτεται. 566. Απορρίπτεται. 567. Απορρίπτεται. 569. Απορρίπτεται. 571. Απορρίπτεται. 573. Απορρίπτεται. 574. Απορρίπτεται. 575. Απορρίπτεται. 5.76 Απορρίπτεται. 5.78 Απορρίπτεται. 6.23 Απορρίπτεται. 581. Άλλος ένας παρακαλώ. Πέρας. Δεκτή.

Απορρίπτεται. 588. Απορρίπτεται. 589. Απορρίπτεται. 590.

Να μην τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Δεν θέλετε. Εξακόσια. Δύο ακόμη, παρακαλώ. Για την 600. Καλώς. Απόλυπτεται. 601. Απορρίπτεται. 603. Απορρίπτεται. 6-12. Απορρίπτεται. 605. Απορρίπτεται. 607 απορρίπτεται 609 απορρίπτεται 611 Απορρίπτεται. 6.13. Απορρίπτεται. 615. Απορρίπτεται. 617. Απορρίπτεται. 6-19. Απορρίπτεται. 40. Απορρίπτεται. 41. Απορρίπτεται. Λοιπόν, επανέλθουμε στις ε, απλές ψηφοφορίες. Διανατάσσου, 42 υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά να την ελέγξουμε. Απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Να την ελέγξουμε λοιπόν. Δεκτή. Ωραία. Σαράντα επτά υπέρ. Κατά. Να την ελέγξουμε. Α, απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ό, ήταν, ήταν σαφές αλλά καλά άμα θέλετε ελέγχουμε τη 48 άλλος ένας απορρίπτεται συμβαστική 16 ηλεκτρονικά Δεκτή. 53 υπέρ. Κατά αποχές. Καλά, εγώ νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά θα θέλετε οπωσδήποτε να ελεγχθεί, οπότε ας ελέγξουμε. Απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 18 ηλεκτρονικά δεκτή 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 19 α συγγνώμη 62 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 19 ηλεκτρονικά. Δεκτή. Συμβαστική 20 ηλεκτρονικά. Δεκτή. 69 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε την 69. Μέχρι και ΙΜΚΟ 3 όλες αυτές. Απορρίπτονται ως συνήθως. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 76 76 απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή α, ελέγχουμε την 79 Δεκτή. Ήμκο 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 22 ηλεκτρονικά. Δεκτή. 88 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήμκο 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήμκο 7 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την Ήμκο 7 Απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ κατά λοιπόν να ελέγξουμε την 95 απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 6 υπέρ όχι συγγνώμη ΙΜΚΟ 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές δεκτή α την ελέγχουμε την 103 δεκτή 104 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε την Ήμκο 9. Απορρίπτεται. 107 και τραν 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Θα έλεγα. Αλλά παρόλα αυτά να ελέγξουμε. Ναι. Δεκτές. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται Συμ... όχι 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 23 ηλεκτρονικά δεκτή συμβαστική 23. Τέσσερα λέει ο πρόεδρος. Δεκτή. Συμβαστική 25. Δεκτή. Συμβαστική 26. Ηλεκτρονικά. Δεκτή. 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τραν 7 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. Συμβαστική 27 ηλεκτρονικά. Δεκτή. Συμβαστική 29 ηλεκτρονικά. Δεκτή. 147 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήμκο 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 30 ηλεκτρονικά Δεκτή. 153 υπέρ. Κατά. Την ελέγχουμε. Την 153. Απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 και ΙΜΚΟ 16 υπέρ κατά αποχές δεκτές συμβαστική 33 ηλεκτρονικά δεκτές 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά απορρίπτεται 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήμκο 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τραν 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 35 ηλεκτρονικά δεκτή 168 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 36 ηλεκτρονικά δεκτή 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 38 ηλεκτρονικά άλλη μια ψήφος όχι δεκτή οπότε 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 181 υπέρ κατά να την ελέγξουμε Απορρίπτεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 40 ηλεκτρονικά. Δεκτή. 186 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 186. Δεκτή. 189 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 190 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 192 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές δεκτή 195 υπέρ κατά ελέγχουμε την 195 απορρίπτεται 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 κατά πρέπει να ελέγξουμε την 197 Α, απερίφθη, 199 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Την έκθεση συνολικά ηλεκτρονικά. Δεκτή. Την απόφαση έναρξης διαπραγματεύσεων. Ο εισηγητής θέλει το λόγο. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω τους κοιόδης που πραγματικά επέδειξαν πολύ θετική διάθεση διαλόγου. Εργαστήκαμε σε ένα επικοδομητικό κλίμα και ευχαριστώ και τη συνεργάτητά μου Τατιάνα Κουμπριά που έκανε πολλή δουλειά και τη γραμματεία της Επιτροπής μας. Νομίζω ότι αυτό που επιτύχαμε σήμερα είναι ένα πρώτο αποφασιστικό βήμα υπέρ μιας καλύτερης προστασίας των καταναλωτών. Τώρα για την εντολή. Ξέρω ότι το Συμβούλιο και η προσεχής Ρουμανική Προεδρία δεν θα είναι έτοιμη πριν από τον Μάιο. Οπότε προτείνω να μην ψηφίσουμε την εντολή σήμερα για να εξακολουθήσουμε να έχουμε την πρωτοβουλία εδώ εμείς στο Κοινοβούλιο και για να έχουμε την καλύτερη, δυνατή και ενοποιημένη θέση ε, εμείς ως Κοινοβούλιο πριν από τις ευρωεκλογές. Γι' αυτό προτείνω να μην ψηφίσουμε επί της εντολής σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το ηθοτήσουμε σε πρώτη ανάγνωση πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές και μπορεί με αυτόν τον τρόπο το Κοινοβούλιο να έχει μία ενιαία θέση και να μπορέσει να έχει περιθώριο επιλογής όσο δεν έχει αποφασίσει το Συμβούλιο. Κυρία Ντεροζιέρ. Δηλαδή, ουσιαστικά αναβάλουμε την ε, εκλογή για την εντολή ή πάει στην Ολομέλεια για έγκριση στην πρώτη ανάγνωση. Πάμε στην Ολομέλεια για πρώτη ανάγνωση, δεν ψηφίζουμε σήμερα την εντολή, δεν ξεκινάει ο τριμερής διάλογος, διότι δεν θα είναι έτοιμο το Συμβούλιο έτσι κι αλλιώς με αυτό τον τρόπο σταθεροποιείται και, και αποκτά το Κοινοβούλιο μια ενιαία θέση πριν το τέλος της θητείας. Εγώ θεωρώ ότι ήταν δύσκολη η επίτευξη συμβιβασμού. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα κείμενο που έχει εγκριθεί στην Επιτροπή. Δεν είμαι λοιπόν υπέρ του να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια πρέπει να παραμείνει το κείμενο όσο έχει και να ξεκινήσει διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Εγώ θα ήθελα να ψηφίσουμε εντολή τώρα. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο κίνδυνος είναι να μην υπάρξει κείμενο μέχρι το τέλος της θητείας μας. Κινδυνεύουμε δηλαδή να χάσουμε τη δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να έχει καλύτερη προστασία προς τους καταναλωτές. Γι' αυτό και δεν θέλω να ψηφίσουμε σήμερα την εντολή. Κρατάμε αυτή τη δυνατότητα δράσης, αν θέλετε, στο Κοινοβούλιο. Αν ξεκινήσουμε τώρα τον τριμερή διάλογο, η επόμενη Προεδρία, η Ρουμανική, μπορεί να μην θέλει να επεξεργαστεί το θέμα. Και εγώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές φήμες για το θέμα αυτό. Δεν θέλω να δώσουμε μήνυμα στο Συμβούλιο ότι δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις. Καλό θα ήταν να συνεχίσουμε τις πιέσεις προς το Συμβούλιο. Είμαστε διατεθειμένοι και έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Εάν σε δύο ή τρεις μήνες δούμε ότι δεν ξεκινάει τίποτα, τότε μπορούμε να πάμε στην Ολομέλεια. Α στείλουμε λοιπόν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο Συμβούλιο και στον Ευρωπαίο Καταναλωτή ότι θέλουμε το συντομότερο δυνατόν να βελτιώσουμε την προστασία τους και να τους δώσουμε περαιτέρω δυνατότητες και μέσα προστασίας. Δεν θα ήθελα αυτό να ερμηνευθεί διαφορετικά με την έννοια ότι δεν θα κινηθεί το Συμβούλιο, γι' αυτό και δεν κάνουμε κι εμείς τίποτα. Ας διατηρήσουμε την πίεση και έχουμε πάντα τη δυνατότητα σε δύο ή τρεις μήνες να πάμε στην Ολομέλεια. Πρόεδρος. Ναι, η Προεδρία χτες με ενημέρωσε ότι δεν θα είναι έτοιμη πριν το Μάιο. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία, πρέπει να ψηφίσουμε αν ναι ή όχι θέλουμε να ψηφίσουμε την, την εντολή. Η κυρία Ροζιέρ. Εγώ ήθελα να συμφωνήσω με την Μάντι Πραγματικά είμαστε ε, αρμόδια αρχή, συναρμόδια για την νομοθεσία εδώ και ουσιαστικά βασιζόμαστε σε φήμες, σε πράγματα τα οποία δεν είναι σίγουρα. Είμαστε συναρμόδια αρχή νομοθετική και δεν καταλαβαίνω από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η θητεία έχουμε ακόμα χρόνο να δράσουμε. Εάν διαπιστώσουμε ότι δεν ανταποκρίνεται το Συμβούλιο, μπορούμε να αλλάξουμε πρακτική. Αυτή τη στιγμή όμως γιατί εμείς να πάρουμε μία απόφαση βάσει πιθανών ε, στάσεων του Συμβουλίου. Πρόεδρος. Υπάρχει η πρόταση να μην ψηφίσουμε. Θα γίνει λοιπόν τώρα μία ψηφοφορία, αν ναι ή όχι θα ψηφίσουμε την εντολή. Συμφωνώ, ε, καταλάβατε όλοι περί τίνος ψηφίζουμε. Ναι, το ερώτημα είναι αν ναι ή όχι θα ψηφίσουμε και ψηφίζουμε γι' αυτό. Καταλάβατε όλοι γιατί ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ του να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Υπάρχει σαφής πλειοψηφία υπέρ του να ψηφίσουμε την εντολή. Για την εντολή. Ψηφίζουμε λοιπόν. Αρχή της ψηφοφορίας. Ε, is adopted. So, anyway, congratulations to Συγχαρητήρια παρόλα αυτά στον εισηγητή. Και θα συνεχίσουμε με την επόμενη ψηφοφορία που είναι η θέση του κυρίου Βέλουκαν αφορά το σχέδιο τροποποίησης του πρωτοκόλου περιοργανισμού του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύκο 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αύκο 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αύκο 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία Τσαμπάσκι. Θα ψηφίσουμε ξεχωριστά υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 τμήμα 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα 2 καταπίπτει. 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 καταπίπτει αύκο 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά ελέγχουμε το 4 Ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται, δεν βλέπω χέρια. Έλεγχος. Εγκρίνεται. Το σύνολο της έκθεσης ψηφίζουμε. εγκρίνεται. Απόφαση για την αρχή των διαπραγματεύσεων. Δεν υπάρχουν εδώ αντιρρήσεις. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Βέλκεν, τον εισηγητή. Και το επόμενο σημείο είναι η ψηφοφορία, μάλλον η έγκριση εντολής των ψηφιακών εργαλείων, αρχή της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τέλος. Την κυρία χάνιβόλα έχουμε την έκθεση μάλλον τέσσερι ψηφοφορίε όσον αφορά τι αστικέ πτυχέ των διεθνών απαγωγών παιδιών. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά πρώτη ψηφοφορία αρχή. Εγκρίνεται. Δεύτερη, 15. γίνεται. 16. Εγκρίνεται. 17. Τέλος. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Κυρία Χάνιμπολ. Ολοκληρώσαμε τις τροπολογίες και θα συνεχίσουμε με τα επόμενα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με το σημείο 18. Θα ήθελα παρακαλώ να σας ζητήσω λίγη ησυχία στο, στην αίθουσα. Το επόμενο σημείο είναι η ενημέρωση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που αφορούν την ε, γνωμοδότηση της κυρίας Νίμπλερ που αφορά το πλαίσιο προληπτικής αναδιάρθρωσης, δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα όσον αφορά διαδικασίες που αφορούν αναδιάρθρωση, αφαιρεγγιότητα και απαλλαγή. Η κυρία Νίμπλερ δεν είναι παρούσα μου ζήτησε λοιπόν να, σα να σας παρουσιάσω αυτά που έχουν συμβεί στον, τριμερί... στον τρίτο διάλογο, τριμερή διάλογο που έγινε την προηγούμενη πέμπτη. Η διαπραγματευτική ομάδα στηρίχθηκε από την σαφή αλλαγή στάσης του Συμβουλίου που έδειξε πρόθεση συμβιβασμού συμβεβασμό απαραίτητου για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Κάποια θέματα που αφορούν την εξισορρόπηση των δικαιωμάτων καθώς και την προάσπιση και εξασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η κυρία Νίμπλερ πιστεύει ότι θα ληφθούν υπόψη αυτά τα σημεία και θα μπορέσει στην επόμενη Ολομέλεια να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για το θέμα αυτό. Υπάρχουν σχόλια? Δεν βλέπω κάποιον. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε με το 19. Ουσιαστικά αφορά τις συμβάσεις ε, για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Από τους συζητητές είναι παρόν μόνο ο κύριος Φως. Έχετε το λόγο. Πρόκειται για τις συμβάσεις, για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ ξεκίνησε ο τριμερής διάλογος. Την τελευταία φορά δεν προχώρησαν ε, και πολύ τα πράγματα. Δεν έχω λοιπόν και πολλά να σας ε, ενημερώσω. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των λεγόμενων smart goods και υπάρχει και μία οδηγία για τα για τα λεγόμενα tangible goods, την οδηγία αυτή, στην οποία θέλουμε να υλικά ψηφιακά. Και ουσιαστικά θέλουμε να δούμε περαιτέρω ε, το βαθμό της εναρμόνισης. Και βεβαίως ε, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη προθεσμία όσον αφορά το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να σας πω και πολλά, παραμένουν δύο ερωτήματα ανοιχτά. Το θέμα της ε, ενημέρωσης αλλά τίποτα παραπάνω ουσιαστικά από την τελευταία φορά που συζήτησαμε για το θέμα αυτό δεν έχω να σας πω. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σχόλια από άλλα μέλη της Επιτροπής, δεν βλέπω κανέναν. Να συνεχίσουμε με το 20. Και άλλη μια φορά πρόκειται για τις διαπραγματεύσεις κανόνες σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων. Εγώ θα σας μιλήσω εκ μέρους των ε, εισηγητών. Την προηγούμενη Τετάρτη, στις 28 Νοεμβρίου, έλαβε χώρα η τελευταία τριμερής ε, συνάντηση, τριμερούς διαλόγου. Σημαντικά πολιτικά θέματα παραμένουν όσον αφορά το θέμα του ορισμού της χώρας προέλευσης, το θέμα της ε, εφαρμογής, το θέμα της μεταβατικής περίοδου, των, ε, της ρήτρα αναθεώρησης και της προθεσμίας ημερομηνίας μεταφοράς. Και βεβαίως όσον αφορά εδώ τα υπόλοιπα θέματα που αφορά την ε, μεταφορά, το θέμα του αν θα υπάρξει κανονισμός από την οδηγία, το θέμα της διεύρυνσης του ορισμού της χώρας προέλευσης παραμένει ακόμα ανοιχτό. Η αναδιατύπωση του άρθρου 2 της αιτιολογικής σκέψης 9β έλαβε χώρα στην πέμπτη συνάντηση τριμερούς διαλόγους και πρέπει να σας πω ότι είναι κοντά τα θεσμικά όργανα σε μια συμφωνία. Χρειάζεται ακόμα λίγη δουλειά έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα κοινά αποδεκτό κείμενο. Θα υπάρξει νέα συνάντηση στις 13 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο και θα συμπεριληφθούν αυτά τα δύο εκρεμή σημεία και προσβλέπουμε στην επίλυσή τους. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό, δεν βλέπω κανέναν. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 21 λοιπόν, που αφορά το θέμα της ε, οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο κύριος Φως. Υπήρξε μια πάρα πολύ μακρά συνεδρίαση στη τελευταία συνάντηση του τριμερούς διαλόγου και το αποτέλεσμα ήταν καλό. Τα πιο σημαντικά σημεία Παραμένουν βέβαια ακόμα ανοιχτά το θέμα της ε, αποθήκευσης δεδομένων, data mining. Το θέμα των δικαιωμάτων ε, των εκδοτών υπάρχει, αν θέλετε, σύγκληση σε κάποια σημεία για το θέμα του value gap, παραδείγματος χάρη, μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου συγκλίναμε λίγο στα σημεία στα οποία ουσιαστικά επικαλυστήκαμε διαφορετικές οδηγίες, διαφορετικά νομοθετικά κείμενα. Η Επιτροπή επιθυμεί να αναπτύξει νέο νομοθετικό κείμενο αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να συγκλίνουμε λίγο. Συζητήσαμε και για κάποια άλλα εκρεμή θέματα, άρθρο 14, 15, που αφορά διαφάνεια, διαδικασίες για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των ε, συγγραφέων και των ε, προεχόντων, τα δικαιώματα. Και εδώ, και εδώ χρειάζεται να πλησιάσουμε οι θέσεις των μεν ή μεν τον λίγο περισσότερο, έγιναν βήματα, το άρθρο 9α τώρα του Συμβουλίου που έχει προσθέσει κάτι, κάτι που δεν είχαμε στο 7-1 Εκεί μπορέσαμε να πετύχουμε μια συμφωνία. Την επόμενη πέμπτη θα λάβει χώρα η επόμενη συνεδρίαση του τριμερούς διαλόγου και συνεχίζουν αν θέλετε, να παραμένουν ανοιχτά οι βασικές δυσκολίες που είχαμε από την αρχή. Ελπίζω, ελπίζω να καταφέρουμε να τα ξεπεράσουμε. Πρόεδρος δεν βλέπω να ζητάει κάποιος το λόγο από τα λίγα μέλη που έχουν παραμείνει στην Επιτροπή, στην αίθουσα. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε την συνεδρίασή μας. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο και θα αρχίσει στις 9 και 4 το βράδυ. Θα είναι βραδινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ.